So, colleagues, I think Πρέπει να ξεκινήσουμε, συνάδελφοι. Μικέλε, γεια σου. Θα περάσω στα, στη μητρική μου γλώσσα. Θα συνεχίσουμε τώρα την συνεδρίαση της Επιτροπής που διακόψαμε στις 12.30. Έχουμε φτάσει στο σημείο 12.30 της ημερήσιας διάταξης ε, που είναι ανταλλαγή απόψεων με το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Ε, χαιρετίζουμε σήμερα εδώ, καλωσορίζουμε τον ε, Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Λιμ, καθώς ε, και τον Διευθυντή του Τμήματος για το Περιβάλλον, τον κύριο Γιαμάντα. Κύριε Λιμ, κύριε Γιαμάντα, σας ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεστε εδώ μαζί μας σήμερα. Μας ε, ακούτε? Ωραία. Η ε, Επιτροπή Τουρισμού σας ευχαριστεί, ε, Μεταφορών και Τουρισμού σας ευχαριστεί για τον χρόνο που μας αφιερώνετε. όσον αφορά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και το περιβάλλον, ε, ο Διεθνής Δευτεριακός Οργανισμός ε, βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής και γι' αυτό θα πρέπει όλοι οι τρόποι μεταφοράς ε, να συμμετάσχουν στην προσπάθεια μείωσης των εκπομπών. Θέλουμε να τεθούν στόχοι όσον αφορά τις εκπομπές, ωστόσο θα πρέπει όλοι οι οικονομικοί φορείς να ε, ακολουθούν ε, τους ίδιους κανόνες. Πιστεύουμε λοιπόν ότι υπάρχουν κάποιες στοιχείες που πρέπει να ληφθούν ε, υπόψη στην όλη συζήτηση. Η συνεργασία ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα την Επιτροπή Μεταφορών και τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό θα πρέπει να ενισχυθούν. Ε, θα δώσω τώρα το λόγο σε εσά ε, για 15 λεπτά και κατόπιν ε, θα δώσουμε το λόγο σε ευρωβουλευτές. Περίπου 5 λεπτά θα μιλήσει ο κύριος Σελίμ και ο κύριος Γιαμάντα θα έχει 10 λεπτά στη διάθεσή του για την παρουσίασή του. Κύριε Ελίμ, παρακαλώ έχετε το λόγο. Uh, thank you, uh, Mr. Chair. Πρόεδρε. Μου δώσατε πέντε λεφτά. Εγώ θα ήθελα να δωρήσω στους ε, συναδέλφους, στους βουλευτές δηλαδή, περισσότερα, περισσότερο χρόνο, γι' αυτό θα μιλήσω μόνο τρία λεφτά. Μεγάλη μου τιμή που με καλέσατε για να σας συναντήσω και σας ε, συγχαίρω για την εκλογή ή επανεκλογή σας. Εκφράζω την εκτίμησή μου για τον επικοδομητικό διάλογο μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας τα τελευταία χρόνια. Προσβλέπω σε περαιτέρω στενή συνεργασία. Ο διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας έχει ασχοληθεί με διάφορα θέματα ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος. Ασχολείται κυρίως όμως με περιβαλλοντικά θέματα ε, και θέματα κλιματικής αλλαγής, γιατί αποτελούν μεγάλη πρόκληση και είναι ψηλά στην ατζέντα του οργανισμού μας. Και ελπίζω να συνεργαστώ πολύ καλά με τους ευρωβουλευτές. Έχουμε 174 συμβαλόμενα κράτη. Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι η πρόοδος που έχουμε σημειώσει δεν είναι ταχεία. Αλλά όλα τα κράτη προσπαθούν να κάνουν προσπάθειες για να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις. Για τα κλιματικά θέματα, ε, μας απασχολεί το τεχνικό επίπεδο, η, αποδοτικότητα των ε, κινητήρων και από την άλλη η βελτιστοποίηση ε, της ταχύτητας. Και επίσης τι θα κάνουμε στο μέλλον με τα καύσιμα για την ε, κίνηση των πλοίων στον τομέα της ενέργειας δηλαδή. Μας απασχολεί και αυτός ο τομέας που είναι σημαντικός. Συνεργαζόμαστε φυσικά για αυτά τα θέματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί έχουμε τους ίδιους στόχους. Πρέπει να συνεργαστούμε μεταξύ μας. Και εγώ κάνω ό,τι μπορώ για να διευκολύνω αυτή την συνεργασία για να αντιμετωπίσουμε διάφορα περιβαλλοντικά θέματα, ειδικά να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή. Αυτά τα θέματα έχουν και ανθρωπιστική διάσταση. Προσπαθούμε να αναπτύξουμε ένα δόγμα, μια φιλοσοφία, όσο μπορούμε, για να μας βοηθήσει να σημειώσουμε πρόοδο. Θα ήθελα λοιπόν να καλέσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεργαστεί και να συνεχίσει να στηρίζει τον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας και εμείς από πλευράς μας θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ούτω ώστε να διατηρήσουμε ψηλά τα πρότυπα και να υπάρχει ισοτιμία μεταξύ όλων. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Λιμ για την εισαγωγή σας αυτή. Θα θέλαμε τώρα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Γιαμάντα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα παρουσιάσω λίγο πιο λεπτομεριακά τα θέματα, αλλά φυσικά με συντομία. Ο IMO είναι εξειδικευμένος οργανισμός του ΟΗΕ για την θαλάσσιες μεταφορές, την ασφάλεια των θαλασσιών μεταφορών και έχει αναπτύξει πάνω από 50 διεθνή κείμενα ανάμεσα σε αυτά το, η Σόλας, η Σύμβαση για την Ασφάλεια στη Θάλασσα και άλλα πολύ σημαντικά. Η... Ε, αναμένουμε μια τροποποίηση σε 1,5 χρόνο εξαιτία φυσικά τη ε, ειδική διαδικασία που ακολουθείται για την τροποποίηση των συμβάσεων του IMO. Έτσι λειτουργούν τα πράγματα σε αυτόν τον οργανισμό. Και το ανώτατο αποφασιστικό όργανο είναι η Γενική Συνέλευση ε, με 134 ε, χώρες που συμμετέχουν σε αυτή. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μια φορά στα τρία χρόνια. Γι' αυτό είναι, πολύ σημαντικό και η λειτουργία του Συμβουλίου, το οποίο συναντάται δύο φορές το χρόνο, έχει 40 ε, κράτη-μέλη, 10 εκ των οποίων είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια ισχυρή φωνή στον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας. Θα ήθελα τώρα να μιλήσω για την ε, σύμβαση Μάρπολ, η οποία είναι η σύμβαση που αναφέρεται στην προφύλαξη των θάλασσών από οποιαδήποτε μορφή ρήπανση από τα πλοία. Για παράδειγμα, πετρελαιοκυλίδες, ε, απορρίψη χημικών ε, ουσιών επικινδύνων ή επίσης τα απορρίμματα, ιδιαίτερα για τα απορρίμματα που περιγράφονται στο παράρτημα 5 της Σύμβασης Μάρπολ, ε, έχουμε ρυθμίσεις πιο συγκεκριμένα και για τα πλαστικά στο παράρτημα 5. Και επειδή έχουμε να ενισχύσουμε την ε, ρύθμιση αυτού του θέματος. Τώρα, εγώ θα ήθελα να αυτοαφερθώ πιο συγκεκριμένα στο παράρτημα της Μάρπολ που αναφέρεται στην ατμοσφαιρική ρήπανση που προκαλούν τα πλοία. Ε, είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό. Θα γνωρίζετε ότι έχουμε τη στρατηγική IMO 2020 για την μείωση των εκπομπών θείου. Να μειωθεί σε 0,5% από το προηγούμενο όριο που ήταν 3,5%. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα που αναλαμβάνουμε και θα έχετε διακούσει ότι ήδη από την 1η Μαρτίου έχει απαγορευτεί η χρήση καυσίμων που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε θείο άλλες προσπάθειες έχουμε αναλάβει για τη μείωση των εκπομπών των οξυδίων του αζότου. Ε, έχουν επίσης ε, εισαχθεί υποχρεωτικές, υποχρεωτικοί δείκτες ενεργειακής αποτελεσματικότητας για τα πλοία και ε, συμπεριλαμβάνονται και οι εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα σε αυτές. Όπως γνωρίζετε, με βάση την αρχική μας στρατηγική ε, προσπαθούμε να ε, επιταχύνουμε την υιοθέτηση αυτών των μέτρων. Στην συνέλευση του Απριλίου ε, προβλέπεται ότι θα ε, υπάρξουν αποφάσεις που θα επιταχύνουν την τρίτη φάση, τη λεγόμενη, δηλαδή ως το 2022 να επιτύχουμε ε, αυτή τη μείωση Βλέπετε εδώ πώς έχει εξελιχθεί το επίπεδο φιλοδοξίας, αν θέλετε, πόσο ε, έχουμε εντείνει τις προσπάθειές μας. Ο στόχος είναι έως το 2030 να υπάρχει μια μείωση 40%. των αερίων του θερμοκηπίου από, από όλα τα πλοία και να επιτύχουμε μια μείωση ε, συνολική 50% μέχρι το 2050 και της έντασης 70%. Ο γενικότερος στόχος είναι να μειωθούν στο μισό μέχρι το 2050 οι εκπομπές σε σχέση με το 2008. Βλέπετε με την μπλε γραμμή στο διάγραμμα θα συμβεί αν συνεχίσουμε ως ήθιστε με την πεπατημένη και δεν αναλάβουμε κάποια πρωτοβουλία και τελικό στόχος είναι μέσα στον αιώνα, τον 21ο, να, μην υπάρχουν, να υπάρχουν μηδενικές εκπομπές από τα πλοία. Και σε αυτό το διάγραμμα βλέπετε τους στόχους της αρχικής στρατηγικής. Σε τη στιγμή έχουμε εκπομπές περίπου 950 εκατομμυρίων τόνων. Στόχος είναι να πέσουμε κάτω από τους 450 μέχρι το 2050 με την πράσινη γραμμή. Το μπλε σκέλος στο διάγραμμα δείχνει τι θα συμβεί αν συνεχίσουμε χωρίς καμία προσπάθεια, αλλά ε, βλέπετε ότι εάν εισαχθούν τα διάφορα τεχνολογικά μέτρα, δηλαδή βελτίωση στα, στα καύσιμα ή στα συστήματα πρόθεσης των πλοίων, θα καταφέρουμε ε, να πετύχουμε αυτό που είναι με πράσινο στο διάγραμμα. Ε, υπάρχουν επίσης και κάποια ε, επιχειρησιακά μέτρα που μπορεί να λάβει κανείς, λειτουργικά μέτρα, όπως για παράδειγμα να εισέρχεται το πλοίο στο λιμένα όταν ακριβώς χρειάζεται, όχι πριν, ή να ευελτιστοποιείται η ταχύτητα του πλοίου. Και αυτά είναι με πορτοκαλί. Εάν μεγαλύτερη υιοθέτηση των καυσίμων, ε, για παράδειγμα βασίζονται στην αμμονία ή στο υδρογόνο, αυτά έχουν μηδενικές εκπομπές. Εάν συ, συ, ε, υπάρξει χρήση όλων αυτών των μέτρων μαζί, πιστεύουμε ότι μέχρι το 2050 θα επιτύχουμε τους στόχους μας. Ένας ακόμα τρόπος να επιτύχουμε τον στόχο των μηδενικών εκπομπών, είναι φυσικά ο IMO ένας παγκόσμιος ρυθμιστικός οργανισμός. Ένας λοιπόν επιπλέον τρόπος είναι να προωθήσουμε την έρευνα και την ανάπτυξη νέων καινοτόμων καυσίμων. Το επιδιώκουμε αυτό σε συνεργασία με κέντρα έρευνας. Επιθυμούμε ο οργανισμός μας να λειτουργήσει ως καταλήτης στην έρευνα που γίνεται παγκοσμίω για την ανάπτυξη νέων μορφών καυσίμου που δεν, έχουν, που δεν προκαλούν εκπομπές. Φαίνεται ότι θα χρειαστούμε έναν μηχανισμό με συμμετοχή τη αγορά. που θα πρέπει να υποστηρίξει αυτές τις νέες τεχνολογίες μηδενικών εκπομπών και καυσίμων μηδενικών εκπομπών. Και εμείς επιδιώκουμε να το υποστηρίξουμε αυτό με με ρυθμίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, οποιαδήποτε πρωτοβουλία από δική σα πλευρά ε, συνεισφέρει είναι προσδεκτή. Βεβαίως, αυτή τη στιγμή εστιάζουμε σε κάποια πιο βραχυπρόθεσμα μέτρα για να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε στο 2050. Όμως παράλληλα, οποιαδήποτε άλλη πρόταση ή ιδέα που μπορεί να εμπλέκει οι παράγοντες της αγοράς είναι χρήσιμη. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να αναλάβουμε δραστηριότητες για να μην μείνει κανείς πίσω, να έχουμε τεχνική συνεργασία, ε, Έχουμε αναπτύξει λοιπόν τέτοιες ε, πρωτοβουλίες, για παράδειγμα ε, δωρεές προς κράτη που χρειάζονται τέτοια τεχνική συνεργασία. Ιδιαίτερα θα ήθελα να αφαιρθώ στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνεργασία για τι Τελάσσιε μεταφορέ ε, και τη δημιουργία κέντρων συνεργασία που έχει χρηματοδοτήσει. Αυτό είναι κάτι που το εκτιμούμε ιδιαίτερο ως πρωτοβουλία, όμως ξέρετε ότι ολοκληρώνεται το πρόγραμμα στο τέλος του 2020. Ε, ο IMO εκτιμά ιδιαίτερο την συνεργασία που, έχουμε, που είχαμε μέχρι τώρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί. Επίσης, η λεγόμενη αρχική στρατηγική προσπαθεί να δώσει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στη βιομηχανία, στον κλάδο, ότι πρέπει και εκείνοι να αναλάβουν πρωτοβουλίες για να πετύχει τις μηδενικές εκπομπές του κλάδου της ναυτιλίας. Συμπερασματικά, θα έλεγα ότι στον IMO ακολουθούμε τη στρατηγική μας και προοδεύουμε πάνω σε αυτήν. Ε, θα υπάρξει μια πρώτη αναθεώρηση του 2023 Είπα ότι θα ενταθούν και οι επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη. Εάν λοιπόν συνδυάσουμε όλες αυτές τις προσπάθειες σε ένα κοινό διεθνές ρυθμιστικό πλαίσιο, μπορούμε να τα καταφέρουμε και ε, προσβλέπουμε στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γιαμάντα, σας ευχαριστώ κύριε για τι εισηγήσει σας εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο Συνήθως ε, δίνουμε το λόγο πρώτα στους ε, συντονιστέ ε, των πολιτικών ομάδων για να θέσουν ερωτήσεις. Και γι' αυτό θα ξεκινήσουμε από το ΕΛΚ. Η Μπάρμπαρα Τάλερ έχει δώσει τη σειρά της στην κυρία Αντάμοβιτς. Κυρία Αντάμοβιτς, σας δίνω το λόγο. Τρία λεπτά δίνουμε στον κάθε ομιλητή. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι τιμή και χαρά μας το ότι βρίσκεστε εδώ σήμερα στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εγώ είμαι νέα ευρωβουλευτής, ε, είμαι νομικός, ε, έχω εργαστεί στο Πανεπιστήμιο ε, του Κτάνσκ, όπου έχουμε τμήμα για το δίκαιο της θάλασσας. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η σημερινή συνάντηση και συζήτηση. Εάν δεν έχετε αντίρρηση θα μιλήσω πολωνικά. Δεν έχω αμφιβολία ότι μία από τις ε, σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε όλοι μας σήμερα είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος. Λαμβάνοντας ε, υπόψη τους ε, τεράστιους όγκους ορυκτών καυσίμων που χρησιμοποιούνται, βλέπουμε σημαντικές εκπομπές ε, και αυτό συμβάλλει ακόμη περισσότερο στην αλλαγή του κλίματος. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει υιοθετήσει μια στρατηγική για σταδιακή μείωση των εκπομπών από τις θαλάσσιες μεταφορές. Το πρώτο στάδιο της στρατηγικής αυτής ήταν η υιοθέτηση ε, το 2015 μαζί με έναν κανονισμό για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την επαλήθευση των ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα ε, στις θαλάσσιες μεταφορές. Το Ευρωκοινοβούλιο αυτή τη στιγμή ασχολείται με την αναθεώρηση του κανονισμού αυτού, ώστε βαθμιαία να μπορέσουμε να έχουμε ένα ενωσιακό σύστημα για παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των στοιχείων και να μπορούμε να συμβάλλουμε έτσι σε, ε, στην παγκόσμια συλλογή δεδομένων για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τις εκπομπές των πλοίων. και γνωρίζετε ότι υπάρχουν δύο συστήματα, ένα ευρωπαϊκό και ένα διεθνές. Τα σκάφη που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πληρούν διπλές προϋποθέσεις όσον αφορά την παρακολούθηση και ε, την υποβολή εκθέσεων. Αυτό αυτή η λύση δεν είναι ιδανική για τους οικονομικούς ε, φορείς, αλλά Σαν να μην φτάνει αυτό, τώρα ξεκινάμε τις εργασίες πάνω στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, ώστε η Ευρώπη μέχρι το 2050 να είναι η πρώτη ήπειρος ουδέτερη ως προς το κλίμα. Αυτό είναι ένα σημαντικό και φιλόδοξο σχέδιο, μέρος του οποίου αποτελεί το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών και η εφαρμογή του στις θαλάσσιες μεταφορές. Και σε σχέση με αυτό έχω να σας θέσω τώρα μία ερώτηση. Είναι ένα θέμα στο οποίο ήδη αναφέρθηκε ο κύριος Γιαμάντα. Έχει να κάνει με την απαλλαγή από εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα Έχω όμως δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Με την ε, στρατηγική του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για μείωση των εκπομπών από τον Απρίλιο του 2018, ε, στο σχέδιο αυτό υπήρχε ένας κατάλογος επιπλέον μέτρων για περαιτέρω μείωση των εκπομπών βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων ε, μέτρων και με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια σχετικά με το δικό σας όραμα όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και αερίων του θερμοκηπίου στη διεθνή ναυτιλία και όσον αφορά το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Πιστεύετε ότι υπάρχει ελπίδα να υπάρξει ένα διεθνές τέτοιο σύστημα διότι οι, μεταφορές, οι θαλάσσιες μεταφορές από τη φύση τους είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Το να περιοριστούμε αποκλειστικά στην Ευρώπη θα σημάνει ε, με την κατάσταση των εκπομπών. Εάν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα θα πρέπει αυτό να γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά τη συνεργασία μέχρι τώρα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Τι εμπειρίες έχετε εσείς και κατά τη γνώμη σας τι θα πρέπει να γίνει για να ενισχυθεί η συνεργασία αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. ο κύριος Ντάνιελσον. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Λιμ και τον κύριο Γιαμάντα για τις παρουσιάσεις τους. Ο οικολογικός προσανατολισμός ε, του ναυτιλιακού τομέα είναι πολύ σημαντικός ε, για να έχουμε κοινωνίες ουδέτερες ε, όσον αφορά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Ε, κοιτώ τις σημειώσεις μου. Έχω κάποιες ερωτήσεις που σχετίζονται με τις παρουσιάσεις σας. καταρχάς, όσον αφορά το χάσμα των εκπομπών για το οποίο μιλήσατε και την ε, μείωση που θα πρέπει να γίνει μέσω καινοτομίας ε, νέων καυσίμων και νέων τεχνολογιών. Προβλέπετε εσείς σε κάποια διεθνή, κάποια παγκόσμια πρωτοβουλία για να επιταχυνθεί αυτή η μετάβαση. Να έχουμε έναν φόρο, για παράδειγμα, στα καύσιμα, ο οποίος ε, να δοθεί αποκλειστικά σε έρευνες για νέα καύσιμα. Και μήπως μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες ε, σχετικά με τις πιθανές τεχνολογίες ε, που ε, μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Θα πρέπει μέχρι το 2025 για να πετύχουμε τους στόχους του 2050 θα πρέπει να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε τις νέες τεχνολογίες. Ε, δεν απέχει πολύ το 2025. Και δεύτερον, όσον αφορά τα μέσα που βασίζονται στην αγορά, η πρώτη ερώτηση σχετίζεται με το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Ε, συζητιέται και σύντομα θα υποβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποιες είναι οι απόψει σας πάνω σε αυτό και τι δυνατότητες υπάρχουν στο μέλλον να υπάρξει ένα διεθνέ τέτοιο σύστημα και αν όχι, τι άλλα μέσα που να βασίζονται στην αγορά φαντάζεστε εσείς ότι θα μπορέσουν να υπάρξουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Από το Ρενιού, κάτι παρακαλώ. Thank you very much, uh, Secretary General, and uh, Ευχαριστώ το Γενικό Γραμματέα. Ε, εκπροσωπώ την κυρία Nightingale που δεν μπορούσε να έρθει εδώ. Χαίρομαι που υπάρχει η Παγκόσμια Συμφωνία για μια στρατηγική να περιορίσουμε τις ε, εκπομπές της ναυτιλίας, της ναυσιπλοίας. Πρέπει να υπάρχει παγκόσμια, σε παγκόσμιο επίπεδο ισοτιμία και περιμένω να ακούσω περισσότερες προτάσεις από το Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας για το θέμα αυτό. Έχω λίγα σχόλια και θα ήθελα να ακούσω επ' αυτών τις απόψεις σας. Πρώτον, για τα μέτρα για το θείο που τέθηκαν σε ισχύ φέτος. Υπάρχει ε, μία προσπάθεια από τους ε, πλειοκτήτες ε, να βάλουν στα πλοία ένα κατάλληλο μηχανισμό για να υποδεχθούν αυτά τα νέα καύσιμα. Ε, για τα εναλλακτικά καύσιμα, τι δυνατότητες και πρωτοβουλίες θα προωθήσει ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας, ούτω ώστε να υπάρχει ελευθερία για τον κλάδο να επιλέξουν εναλλακτικά καύσιμα, τα καλύτερα δυνατά. Τέλος. Υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίε για καινοτομία, ούτω ώστε να μειώσουμε το αποτύπωμα της ναυτιλίας στο περιβάλλον. Έχει ιδέες ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας για να δώσει κίνητρα για αυτές τις πρωτοβουλίες και για να προωθήσει νέε. Ähm, και εγώ θα ήθελα να θέσω κάποια ερώτηση ως Ευρωβουλευτής και εγώ. Από ό,τι κατάλαβα, μάλλον μιλήσατε ως συντονιστής. Θέλετε να θέσετε κι εσείς κάποια ερώτηση δική σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα πάρω τότε πάλι το λόγο. Κύριε Γενική Γραμματέα, πολύ χαίρομαι που βρίσκεστε εδώ σήμερα, διότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Ε, είναι και πολύ καυτό το θέμα εάν η ναυτιλία θα συμπεριληφθεί στο σύστημα εμπορία εκπομπών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι διαφυσβήτητο ότι ο, ο τομέα τη ναυτιλία θα πρέπει να περιορίσει το οικολογικό του αποτύπωμα, όπω μα είπατε κι εσεί ήδη σήμερα. Οι ε, προκλήσει ε, που αφορούν την αλλαγή του κλίματο θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο, θα πρέπει να θυμόμαστε επίση ότι οι προκλήσει αυτέ δεν μπορούν να λυθούν αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να γίνει μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό τα μέτρα που εφαρμόζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορούν να εξαχθούν. Και γι' αυτό προς τον Διεθνή Ναυτο, Ναυτιλιακό Οργανισμό ε, ρωτώ το εξής. Ε, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών δεν ε, μπορεί να εξαχθεί και Δεύτερον, η ναυτιλία ε, αποκλειστικά εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιπροσωπεύει ε, το 17% ε, μόλις των παγκοσμίων εκπομπών και πάνω από το 80% των ε, εκπομπών, αν θέλουμε να το περιορίσουμε, θα πρέπει αυτό να γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο. Γι' αυτό πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βρει τα ε, κατάλληλα μέτρα που να βασίζονται στην αγορά και που να μειώσουν τι ε, εκπομπέ των πλοίων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι δηλαδή μέτρα που να μπορούν να εφαρμοστούν και εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μειώσουμε τις εκπομπές σε παγκόσμιο επίπεδο. Και τέλος, Υπάρχει το γνωστό θέμα της ε, μετεγκατάστασης ε, των ε, εκπομπών. Ένα μονομερές ε, σύστημα λοιπόν ε, θα έπρεπε να το λάβει αυτό υπόψη του. Γι' αυτό το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας εκπομπών ε, δεν είναι το κατάλληλο μέτρο για να περιορίσει τις εκπομπές από την αυτιλία. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Θα ήθελα πολύ να ακούσω τις δικές σας απόψεις σχετικά με την μετακατάσταση των εκπομπών και ένα σύστημα και τον περιορισμό των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα που να μπορεί να λειτουργήσει σε παγκόσμιο επίπεδο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ από τους πράσινους η κυρία Πάουλου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Γενικό Γραμματέα. Ευχαριστώ τον κύριο Γιαμάντο που ήρθε εδώ. Μεγάλη μας τιμή. Που μας διαθέτετε το χρόνο σας για να μας εξηγήσετε τα μέτρα του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας του IMO, το εκτιμούμε. Είμαι η συγγήτρια για τον φάκελο αυτό και θα ήθελα να σκεφτούμε μαζί κάποια πράγματα. Σε ό,τι αφορά την παρουσίασή σας. Στην τελευταία διαφάνεια είπατε ότι είναι σημαντικό να περιορίσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας στον 1,5 βαθμό Κελσίου. Ένα από τα πιο σημαντικά κράτη που συμμετέχουν στον ΑΕΜΟ, στον ΑΕΜΟ ε, τα νησιά Μάρσαλ θα κινδυνεύσουν αν αυξηθούν τα επίπεδα της θάλασσας. Επομένως θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό πώς συνδυάζεται με τις κλιματικές φιλοδοξίες και με τους δικούς σας στόχους. Γιατί είπατε ότι θέλετε να μειώσετε ε, μέχρι το 2050 τις εκπομπές κατά 50%. Ε, διάβασα διάφορες επιστημονικές εκθέσεις πρόσφατα που οι επιστήμονες λένε ότι για να έχουμε 40% δυνατότητα ε, να μειώσουμε την αύξηση θερμοκρασία στον 1,5 βαθμό Κελσίου, θα πρέπει να είμαστε ουδέτεροι ως προς τις εκπομπές το 2040. Επομένως δεν πρέπει να περιμένουμε το 2050 για να μειώσουμε το κατά 50% τις εκπομπές. Πώς θα μπορέσετε να μας δώσετε, να μας εξασφαλίσετε αυτές τις κλιματικές φιλοδοξίες που θέλουμε. Όταν μιλούσαμε με συμφεροντούχους γιατί το έχω κάνει πολύ τους τελευταίους μήνες και εβδομάδες, μου είπαν ότι οι πελάτες τους τους ζητούν να τους πούν ποιο είναι το αποτύπωμα του διοξιδίου του άνθρακα των αγαθών που μεταφέρει ο διεθνής οργανισμός, δηλαδή που μεταφέρονται μέσω ναυτιλιακών, μέσω πλοίων ας πούμε. Και είπαν ότι θα πρέπει να... Φυσικά Όλοι οι πλειοκτήτες ξέρουν αυτά και χρειαζόμαστε ε, κάποια στοιχεία για να, υπολογίσουμε το αποτύπωμα. Θα αναθεωρήσετε τα DCS για να συμπεριληφθεί και αυτός ο, αυτή η παράμετρος, ούτως ώστε να υπάρχει ισοτιμία σε όλο τον ναυτιλιακό κλάδο για το ETS. Μέχρι στιγμής η ναυτιλία είναι ένας από τους λίγους τομείς, όπως και η αεροπορία, που δεν ε, υπόκειται σε τιμολόγηση των αερίων. Και ένα σύστημα τιμολόγηση των αερίων, φόρο, ε, σύστημα ανταλλαγή εκπομπών μπορεί να δώσει έσοδα για την ε, έρευνα και ανάπτυξη ή για, για μικρά πλοία, ας πούμε, ή για εταιρείε που δεν μπορούν να κάνουν τις απαραίτητες επενδύσεις από τα δικά τους κεφάλαια, με ίδιους πόρους δηλαδή. Και όταν το 2023 θα τσεκάρετε την απόφαση καλό θα ήταν να έχουμε ένα προσχέδιο στο, στα χέρια μας και να έχουμε και κάποια εμπειρία με κάποιο σύστημα τελικά. Σωστό δεν είναι αυτό. Και εδώ, για να απαντήσω τον κύριο Γκάλερ, αν στο ETS έχουμε, ή μάλλον αν έχουμε ETS στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα έχουμε ένα τέτοιο σύστημα μόνο για τους Ευρωπαίους ε, πλειοκτήτες. Θα το έχουμε για όλους. Για όλα τα πλοία τα οποία μπαίνουν σε λιμάνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα από τη σημαία τους, ανεξάρτητα από την πλειοκτησία, ανεξάρτητα από το ποιος είναι στο πλοίο. Θα είναι ένα ισότιμο μέτρο. Θα μπορούσαμε να το έχουμε το 2023. Αν έχουμε ένα κλειστό ETS, ειδικά για την ναυτιλία, θα μπορούσαμε να καλέσουμε όλους να συμμετάσχουν και να αναπτυχθεί αυτό το σύστημα, ας πούμε, σε όλο τον κόσμο. Καλό δεν θα ήταν αυτό το βήμα, γιατί η κλιματική κρίση επιταχύνεται. Θα διαβάσατε τα τελευταία νέα για τις εκπομπές μεθανίου, που είναι πολύ ανησυχητικά νέα. Γι' αυτό λοιπόν σας ε, παροτρύνω να προωθήσετε την κλιματική δράση το συντομότερο δυνατό. Δεν βλέπω να ζητάει κανείς άλλο το λόγο. Έχω εγώ μια ερώτηση. μια πρακτικής φύσης ερώτηση. Και στη Γερμανία, στα λιμάνια μας, βλέπουμε κρουαζιερόπλια. Ε, πλοία που χρειάζονται ε, ηλεκτρικό ρεύμα και χρησιμοποιούν τις δικές τους γεννήτριες και αυτό αν ε, φορτίζουν ε, ηλεκτρικό ρεύμα στο λιμάνι, αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ. Είναι δυνατόν ε, να υπάρξει τέτοιος εξοπλισμός σε όλα τα κανάλια και από οικονομικής πλευράς και από διοργανωτικής πλευράς. Σας ευχαριστώ πολύ και περιμένουμε να ακούσουμε τις απαντήσεις σας. Uh, thank you, uh, uh, Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να απαντήσω σε ένα βασικό ερώτημα και μετά θα καλέσω τον ε, Διευθυντή, τον κύριο Γιαμάντα, να απαντήσει στα υπόλοιπα. Καταρχάς, ε, λοιπόν, ε, λόγω της Συμφωνίας του Παρισιού, που υιοθετήθηκε το 2015 που υιοθετήσαμε τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Πριν από αυτά ήταν τελείως διαφορετική κατάσταση, πριν από τη Συμφωνία του Παρισιού και πριν από τους στόχους ε, βιώσιμης ανάπτυξης. Ε, εμένα μου έκανε εντύπωση η αλλαγή που έχει γίνει. Έχουμε 174 κράτη-μέλη και έχει ε, υπάρξει μεγάλη ευαισθητοποίηση στα θέματα αυτά σε σχέση με πριν. Και ένα από τα στοιχεία ε, είναι 10 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να δημιουργηθούν περιφερειακά κέντρα ε, συνεργασίας ε, για την τεχνολογία. Έτσι λοιπόν ε, παρέχεται εκπαίδευση και κατάρτιση πάνω στην αλλαγή του κλίματος ε, στις διάφορες περιφέρειες και αυτό λειτουργήσε τέλεια στην Κίνα, στον Παναμά, στην Κένια. Αυτό λοιπόν έχει λειτουργήσει πολύ καλά και ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός ε, έχει εφαρμόσει διάφορα προγράμματα συνεργασίας. Όλες οι προσπάθειες ε, ε, συνδυάζονται ε, μεταξύ τους με βάση την Συμφωνία του Παρισιού και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Έχουν αλλάξει πολλά λοιπόν. Δεύτερον, υπάρχει μια παρανόηση όσον αφορά τις συνολικές μας φιλοδοξίες. Το 50% μέχρι το 2050 σημαίνει ότι αν σκεφτούμε την ε, αύξηση του στόλου. Εάν κοιτάξουμε το κάθε σκάφος, η απόδοση, η ενεργειακή απόδοση του πλοίου αυτού θα πρέπει να αυξηθεί κατά 80%. Λέμε λοιπόν 50% τουλάχιστον συνολικά για τις εκπομπές ε, μέχρι το 2050, αλλά σε επίπεδο σκάφους αυτό σημαίνει τουλάχιστον 80 τα Είναι τεράστια αυτή η φιλοδοξία. Αυτό λοιπόν είναι το ένα. Όπως ανέφερε ο διευθυντής μας, υπάρχει ένας πολύ σημαντικός παράγοντας ε, απόδοσης των μηχανών. Αυτό μπορεί να καλύψει περίπου το 50% της μείωσης ε, των ε, εκπομπών. Αλλά τι κάνουμε με το υπόλοιπο 50%? Χωρίς ε, κάποια μελλοντική μορφή ενέργειας δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο, το στόχο μας. Γι' αυτό βασιζόμαστε στην έρευνα και ανάπτυξη, στην εξέβρεση νέων καυσίμων για να τα χρησιμοποιήσουμε στον τομέα της ναυτιλίας. Αυτές τις προσπάθειες λοιπόν εντείνουμε αυτή τη στιγμή. Και όσον αφορά το τελευταίο θέμα που ανέφερε ο Πρόεδρος, όσον αφορά την ε, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, για παράδειγμα, στα κρουαζιερόπλια. Είναι ένα θέμα αυτό. Οι διευκολύνσεις που παρέχουν οι διάφοροι λιμένες. Ε, κάποιοι λιμένες ε, έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν ε, γραμμή παροχής ρεύματος στα κουραζιερόπλια, ώστε να μην χρειάζεται να έχουν αναμένες τις γεννήτριές τους. Αλλά είναι περιορισμένος ο αριθμός των λιμένων που παρέχουν την υπηρεσία αυτή. Ευτυχώς πέρσι είχαμε ένα κοινό ψήφισμα μαζί με τον ε, Διεθνή Οργανισμό Λιμένων για να συνεργαστούμε και να ε, μειώσουμε, να περιορίσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Ε, οι λιμένες λοιπόν συνεργάζονται με το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Ε, θα και άλλους λιμένες να παρέχουν τη δυνατότητα αυτή. Θα παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις και θα συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε τους λιμένες να το κάνουν αυτό. Και ένα άλλο πολύ ευαίσθητο θέμα που θίξατε, ε, θα το αφήσω στον ε, Διευθυντή να απαντήσει στο δύσκολο αυτό θέμα. Um, ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Γενική Γραμματέα. Θα έρθω σε κάποια πιο συγκεκριμένα θέματα. Πρώτα απ' όλα, το σύστημα συλλογής ε, δεδομένων και το MRV είναι διαφορετικά συστήματα, πράγματι. Όμως προσπαθούμε να έχουμε όλο το δυνατόν μεγαλύτερη εναρμόνιση. Ιδιαίτερα για παράδειγμα να έχουμε στοιχεία όπως αυτά αναφέρα, που αναφέρεται η ποσότητα του φορτίου που μεταφέρεται. Είναι μια παράμετρος που προσπαθούμε να εντάξουμε στο, στις, αυτές που συλλέγουμε. Συνεχίζουν να υπάρχουν διαφορές, αλλά υπάρχει σύγκληση το σημαντικό βέβαια και για το MRV και για το DCS είναι να έχουμε ε, επικαιροποιημένα δεδομένα τελευταίες, τις τελευταίες στιγμής από τα πλοία. Ε, η χρήση του DCS, του συστήματος συλλογής δεδομένων, έγινε από το 2019 υποχρεωτική, ενώ το MRV συνεχίζει να είναι προαιρετικό πιστεύω ότι με τα δεδομένα που θα συλλέξουμε μέσω του DCS θα έχουμε τη δυνατότητα να τα αναλύσουμε στη Γενική Γραμματεία του Οργανισμού και μετά από δύο-τρία χρόνια που θα τα διαθέτουμε και θα τα έχουμε αναλύσει, θα μπορέσουμε να τα αξιοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα για να αναθεωρήσουμε τη στρατηγική μας. Γιατί όπως σας είπα το 2023 έχει προβλεφθεί η αναθεώρηση. Άρα πιστεύω ότι περίπου το 2022 θα έχουμε κάποια στατιστικά που θα μας βοηθήσουν να αναθεωρήσουμε τη στρατηγική. Ε, από εκεί και πέρα έχουν γίνει μελέτες που κοιτούν προηγούμενες ε, πρωτοβουλίε, μάλλον που κοιτούν τι παλαιότερε εκπομπέ και προσπαθούν να κάνουν πιο προβολέ στο μέλλον. Όλε αυτέ τι μελέτε θα τι συνυπολογίσουμε στην αναθεώρηση τη στρατηγική. Τώρα κάτι ακόμα. Σχετικό επίση. Το σύστημα εκπομπή, το ECTS, και αν αυτό μπορεί να γενικευτεί. Σας ανέφερα ότι η γενική μας ταχυγική στρατηγική αναφέρεται σε μέτρα τα οποία βασίζονται στην αγορά, αλλά αυτά κατηγοριοποιεί ως μεσοπρόθεσμα μέτρα, δηλαδή από το 2023 έως το 2030. Ταυτόχρονα όμω, η στρατηγική προβλέπει ότι ότι οποιαδήποτε πρόταση για ένα μέτρο το οποίο βασίζεται στην αγορά είναι ευπρόσδεκτη και πριν το 2023. Άρα, εάν υποβληθεί μια καλά τεκμηριωμένη πρόταση στην ε, αρμόδια επιτροπή στην MEPC του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας θα μπορούσε να τύχει επεξεργασίας. Όμως αυτό το σύστημα θα πρέπει να είναι παγκόσμιο για οποιοδήποτε ε, μάλλον δεν είναι απαραίτητο να είναι, ε, να είναι παγκόσμια εφαρμογή. Μπορεί κάποιο να δημιουργήσει ένα σύστημα που να βασίζεται στην αγορά και να το εφαρμόσει σε, σε κάποιε περιπτώσει. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου. Όμω, μια και θέτεται το ζήτημα τη μείωση τη αύξηση τη θερμοκρασία κατά 1,5 βαθμό, ε, πράγματι αυτή τη στιγμή η στρατηγική του 2018 βασιζόταν στα συμπεράσματα του Διεθνούς Πάνελ για το Κλίμα, του IPCC, που έθετε τους τρεις βαθμούς ως υποχρεωτικούς και έλεγε ότι μπορούμε εθελοντικά να κάνουμε μεγαλύτερες προσπάθειες. Ε, και πάλι αυτό το ζήτημα θα τεθεί όταν θα έρθει η ώρα της αναθεώρησης της στρατηγική, το 2023 δηλαδή, με βάση τα στοιχεία και τις μελέτες που θα έχουμε συλλέξει ω τότε. Θέλουμε να έχουμε μεγάλο βαθμό φιλοδοξίας. Αυτή τη στιγμή λέμε ότι ο στόχος της πλήρους ε, ε, των μηδενικών εκπομπών είναι για το μέχρι το τέλος του αιώνα. Αλλά μπορεί κατά τη διάρκεια του αιώνα να καταφέρουμε να τον πετύχουμε πιο νωρίς. Βέβαια, ας μην ξεχνούμε ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας είναι ένα παγκόσμιο φόρο που θα πρέπει να λάβει υπόψη του κανείς ε, και το γεγονός ότι υπάρχουν λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Ε, χώρες δηλαδή οι οποίες θα χρειαστούν υποστήριξη σε άλλους τομείς της οικονομίας τους ίσως. Ε, είναι και αυτό ένα μέλημα. Θα Θέλουμε να είμαστε φιλόδοξοι, φροντίζοντας όμως όλους. Υπήρξαν και άλλες ερωτήσεις, πιο συγκεκριμένες. Το ανέφερε ήδη ο Γενικός Γραμματέας, ότι είναι απαραίτητο να γίνει έρευνα και ανάπτυξη για καύσιμα νέα γενιά που να μην προκαλούν εκπομπέ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πιστεύω ότι στην επόμενη συνάντηση τη MEPC τον Απρίλιο θα εξετάσουμε προτάσει που έχει υποβάλει η βιομηχανία και πιο συγκεκριμένα η AIMRB, ε, το Διεθνέ Συμβούλιο Έρευνα στον τομέα τη ναυτιλίας, το οποίο μας έχει υποβάλει μια πρόταση. Είναι σπάνιο αυτό. Η πρόταση είναι να υπάρξει ένα τέλος υποχρεωτικό που θα επιβληθεί στα καύσιμα και τα έσοδα από αυτό να χρησιμοποιούνται για να γίνει έρευνα για νέες γενιές καυσίμων. Αυτό πιστεύω είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση θα δούμε την εξέλιξη και το αποτέλεσμα της ε, συζήτησης ε, τον Απρίλιο. Κατά πάση πιθανότητα θα συνεχιστεί η συζήτηση και σε επόμενη σύνοδο, δεν θα καταλήξει τον τον Απρίλιο. Έρχεται λοιπόν αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση από την ίδια τη βιομηχανία, αλλά και εμείς από την πλευρά μας έχουμε ξεκινήσει την αξιολόγηση κύκλου ζωής δηλαδή τον υπολογισμό του συνολικού ενεργειακού αποτυπώματος σε όλο τον χρόνο ζωής. Ε, και έχουμε αρχίσει να αναπτύσσουμε σχετικές κατευθυντήριες ε, ε, οδηγίες για το πώς, με ποια μεθοδολογία πρέπει να γίνεται αυτό ανάλογα με το είδος του καυσίμου. Και όπως έλεγα, στο μέλλον θα πρέπει να σκεφτούμε και να αρχίσουμε να υιοθετούμε μέτρα που να βασίζονται στην αγορά. Τώρα, νομίζω για το ETS ήδη μίλησα αρκετά. Θα μείνω εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, thank you, Mr. Ε, Chairperson. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μετά τις απαντήσεις του Διευθυντή μου, θα ήθελα και εγώ να πάρω το λόγο για να προσθέσω κάποια πράγματα, για να μιλήσω λιγάκι για τα μέτρα που βασίζονται στην αγορά και αφορούν το ETS. Έχουμε μέτρα πραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα με βάση τη στρατηγική μας. Ε, τα μέτρα της αγοράς συμπεριλαμβάνονται. Τώρα θέλουμε να αναθεωρήσουμε τη στρατηγική μας μέχρι το 2023 και τα μέτρα της αγοράς συμπεριλαμβάνονται εδώ. Θα μιλήσουμε σε αυτή την αναθεώρηση για αυτά τα μέτρα της αγοράς. Όπως είπαν και οι ευρωβουλευτές, η ναυτιλία είναι ένας παγκόσμιος κλάδος και είναι και πιο περίπλοκη σε σχέση με την αεροπορία. Υπάρχουν θέματα εθνικότητας, οικονομικά θέματα. Είναι πολύ πιο περίπλοκη από την αεροπλοεία, η ναυσιπλοεία. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν παγκόσμια καθολικά πρότυπα για αυτά τα μέτρα αγοράς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σκέφτεται κάποιους μηχανισμούς, όπως το ETS, το μηχανισμό ανταλλαγής ε, εκπομπών. Επίσης, ε, σκοπεύει να κάνει και κάποια μελέτη αντικτύπου γι' αυτό. Όταν η πρότασή της υποβληθεί στον IMO, θα συζητήσουμε τα υπέρ κατά, τι είναι πιο αποτελεσματικό, πόσο συνεισφέρουμε στην μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα για να είναι βιώσιμη η ναυσιπλοεία και θα προτείνουμε ένα παγκόσμιο μηχανισμό. Θέλω να τονίσω ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας παγκόσμιος μηχανισμός. Γιατί αλλιώς θα έχει αρνητικές επιπτώσεις και θα υπάρξει στρέβλωση στον τρόπο που λειτουργεί η ναυσιπλοεία. Επίσης, τα τεχνικά επιχειρησιακά θέματα καλύπτουν μόνο το 50% της μείωσης. Εάν δεν λύσουμε και το θέμα της ενέργειας, των καυσίμων, δεν θα, λύσουμε δεν θα υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Υπάρχουν τεχνολογικές εξελίξεις. Πώς θα τα εφαρμόσουμε στα ποντοπόρα πλοία όμως αυτά τα, νέα στοιχεία ας πούμε. Αν υπάρξει μεγαλύτερη προσπάθεια μπορούν να βρεθούν λύσεις όχι πολύ όχι με πολύ μεγάλο ε, ορίζοντα. Και επίσης θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα στα κράτη που έχουν ε, μεγάλους τόλους να κάνουν επενδύσεις. Έχουμε τα βιοκαύσιμα, την αμμονία, το υδρογόνο. Υπάρχουν τεχνολογικές εξελίξεις εκεί. Αλλά πώς θα τροποποιήσουμε όλες αυτές τις τεχνολογίες που έχουμε για να τις προσαρμόσουμε και να τις εφαρμόσουμε τελικά και στα ποντοπόρα πλοία. Σε ό,τι αφορά την πλυντρίδα, αυτή τη βδομάδα ε, στον IMO δημιουργήθηκε μια υποεπιτροπή για την πρόληψη ε, της ε, ρήπανσης. Και ένα από τα θέματα είναι ακριβώς η πλυντρίδα που καθαρίζει από τα αέρια. Προσπαθούμε να έχουμε κάποια κριτήρια εναρμόνισης για τις ε, εκροές αυτές ε, αερίων από την πλυντρίδα. Θα τελειώσουμε αυτή τη δουλειά μέχρι τα τέλη του επόμενου έτους. ούτως ώστε να χρησιμοποιηθεί και παγκόσμια. Τα θέματα βέβαια είναι τελείως διαφορετικά ανάλογα με το μέγεθος του λιμανιού. Αν είναι μικρό ο κόλπο, ας πούμε, και μικρό το λιμάνι, ε, έχουμε άλλα δεδομένα. Θα επιταχύνουμε τη διαδικασία όσο μπορούμε περισσότερο, ώστε αν γίνεται να έχουμε τα έτοιμα, τα σχετικά μέτρα για την πλυντρίδα, όχι στα τέλη του επόμενου έτου, αλλά στα μέσα. Αυτά ήθελα να πω πέρα από αυτά που είπε ο Διευθυντή μας. Και κάτι άλλο ακόμα. Όταν υιοθετήσαμε τον Οκτώβριο του 2016 την νομοθεσία για το θείο, ήμουν στο πρώτο έτος της θητείας μου. Και η Επιτροπή Προστασίας του Περιβάλλοντος ε, συζήτησε πολύ αυτό το θέμα για το τι θα εφαρμόσει το 20% αν θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τα μέτρα του θείου μέχρι το 2020 ή μέχρι το 2025. Εγώ δεν ήξερα πώς θα το εφαρμόσουμε αυτό, ε, γιατί αφορούσε και την, ε, τα δηληστήρια ε, και την αυσιπλοεία ε, ήταν πολύ συμφεροντούχοι, ήταν πολύ φορείς. Πώς θα μπορούσαμε να συνεννοηθούμε για να εφαρμόσουμε τα νέα μέτρα ε, που αφορούσαν ε, κλάδους που, που δεν κάλυπτε ο IMO. Υπήρχε εξάλλου μεγάλος καυγάς στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Τελικά όμως μέχρι το Φεβρουάριο ε, συνεννοηθήκαμε τότε και πέρασαν απρόσκοπτα τα μέτρα για το θείο. Και εμεί έχουμε φιλοδοξίες και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει φιλοδοξίες. Αν συνεργαστούμε, μπορούμε να βρούμε λύσεις και να τις εφαρμόσουμε μαζί. Εγώ τέλειωσα την πρώτη μου θητεία, την τετραετία μου, και ξεκίνησα ε, τη δεύτερη τετραετία μου, είναι το πρώτο έτος. Έχω συναντηθεί και στο παρελθόν με ευρωβουλευτές, έχουν έρθει στον IMO. Ε, εκτιμώ αυτή τη συνεργασία. Είμαι αισιόδοξο εκφύσεως και πιστεύω ότι χάρη σε αυτή τη συνεργασία μπορούμε να ξεπεράσουμε διάφορα προβλήματα. Αυτά ευχαριστώ. Thank you Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν παρόντες εδώ σήμερα, κύριε Λίμ, κύριε Γιαμάντα. Νομίζω ότι διαπιστώσατε ότι είναι σημαντικό και για τη δική μας Επιτροπή να έχουμε σε τακτική βάση ανταλλαγές μαζί σας. Ξέρω ότι είσαστε σε τακτική βάση προσκεκλημένοι και άλλων επιτροπών του Κοινοβουλίου. Ε, ελπίζω όμως να θεωρείτε και τη δική μας ε, ε, επιτροπή σημαντική και θα ήθελα να σας καλέσω στο όνομα των συναδέρφων μας να μας ξαναεπισκεφτείτε στο μέλλον και μάλιστα να μας επισκέπτεστε σε τακτική βάση. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Ε, ε, περαστικά σας εύχομαι, διότι στο σκι κατάλαβα ότι είχατε κάποιο ατύχημα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ θερμά. Ένα λεπτό διάλειμμα και μετά θα συνεχίσουμε. Thank you very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 Συνάδελφοι, προχωράμε στο επόμενο και τελευταίο θέμα της σημερινής διάταξής μας σήμερα. Θα μιλήσω πάλι γερμανικά. Έχουμε τώρα ανταλλαγή απόψεων ε, με το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ να καλωσορίσω την κυρία Ψέβα, η οποία ε, είναι αναπληρωματική Γενική Διευθύντρια του Κοινού Κέντρου Ερευνών και θα μας παρουσιάσει τις ενέργειες του Κοινού Κέντρου Ερευνών στον τομέα των μεταφορών. Έχει μεγάλη σημασία ε, για την Επιτροπή μας να μάθουμε περισσότερα για τις δραστηριότητες αυτές. Ε, οι νέες τεχνολογίες θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κυρία Βιτσέβα, σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε παρούσα. Ε, θα ήθελα να σας δώσω το λόγο. Περίπου 15 λεπτά έχουμε προβλέψει για την ε, εισηγήσή σας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλό μεσημέρι σε όλους. Πάντα είναι χαρά μου να επισκέφτομαι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι θεωρούμε ότι πρέπει να είμαστε δημοκρατικοί και ανοιχτοί απέναντι στους πολίτες και τους άμεσα εκλεγμένους εκπροσώπους τους. Ε, γι' αυτό είναι μεγάλη χαρά για μας να μπορούμε να σας παρουσιάσουμε τις εργασίες μας. Για όσους από εσά δεν γνωρίζετε το Κοινό Κέντρο Ερευνών, ίσως θα ήταν χρήσιμο σε 30 δευτερόλεπτα να σας εξηγήσω ποιοι είμαστε. Είμαστε η υπηρεσία, η επιστημονική ε, υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 30 ε, τμήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμβουλεύουμε και ε, στόχος μας, ρόλος μας είναι ε, να συγκεντρώνουμε τις γνώσεις που είναι απαραίτητες για τη διαμόρφωση πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με υπερηφάνεια λοιπόν στηρίζουμε με ανεξάρτητες πληροφορίες ε, την λήψη αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε όλον τον κύκλο λήψης αποφάσεων. Βλέπετε λοιπόν εδώ το όνομά μου. Ενημερωτικά σας δείχνω την πρώτη διαφάνεια. Η Επίτροπος η Αρμόδια για μας είναι η Μαρία Γκαπριέλ, ε, που είναι επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης ε, ε, Καινοτομίας και Ερευνών, αλλά και πολιτισμού, εκπαίδευσης και νεολαίας. Και βλέπετε εδώ μια διακεκομένη γραμμή προς τον ε, επίτροπο, τον ε, αντιπρόεδρο για διαθεσμικές ε, σχέσεις, που είναι μάλλον ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για εσάς, επειδή ασχολείται με τις διαθεσμικές σχέσεις, αλλά είναι και αρμόδιος για τις προβλέψεις και την διαμόρφωση πολιτικής. Σε πέντε κράτη κράτη-μέλη εδρεύουμε. Έχουμε έξι εγκαταστάσεις, δύο στο Βέλγιο. Έχουμε το κεντρικό μας γραφείο, αλλά και στο Χέλ, στις κατοχώρες, στην Καρζούη, στη Γερμανία, στην ε, Σεβίλη της Ισπανίας και στην Ιταλία επίσης. Αποστολή μας είναι να παρέχουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποιοτικές ε, και ανεξάρτητες ε, γνώσεις να ε, τροφοδοτούμε δηλαδή τον κύκλο πολιτική με επιστημονικά στοιχεία. Ε, έχουμε πολλές εταιρικέ σχέσεις, ε, διότι όπω κάθε ερευνητικός φορέας χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο αναφοράς. Έχουμε λοιπόν σχέσεις με πολλά ερευνητικά κέντρα σε όλο τον κόσμο. 1.400 επιστημονικές δημοσιεύσεις το χρόνο έχουμε και Είμαστε έτσι ο, ο τρίτος μεγαλύτερος ε, φορέας στον κόσμο όσον αφορά τις ε, παραπομπές που γίνονται ε, σε, δημοσιευ... σε δημοσιεύσεις μας, διότι όταν μιλάμε για αξιοπιστία αυτός είναι πολύ σημαντικός δείκτης. Τι κάνουμε όσον αφορά τις οδικές μεταφορές και τι προκλήσεις μας περιμένουν. Μάλλον θα είναι χρήσιμο καταρχάς να σας δώσω να σας παρουσιάσω τις πιο μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα και στο μέλλον. Οι οδικές μεταφορές δυστυχώς ε, παραμένουν ε, η αιτία για 25.000 θανάτους το χρόνο στην ε, Ευρώπη και ένα εκατομμύριο τραυματίες το χρόνο. Όσον αφορά την οικονομική πτυχή, το 1 με 2% ε, του ΑΕΠ είναι η οικονομική ζημιά λόγω της συμφόρησης στους δρόμους. Ε, και όσον αφορά την ε, πράσινη πτυχή, την οικολογική πτυχή, δυστυχώς οι οδικές μεταφορές παραμένουν ένας από τους σημαντικούς παράγοντες ρήπανσης. Μαζί με τη θέρμανση είναι η βασική αιτία ρήπανση του αέρα, ιδιαίτερα στι αστικέ περιοχέ ε, και είναι και η δεύτερη πηγή ε, αερίων ε, του θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλά προβλήματα λοιπόν εδώ πρέπει να λυθούν όσον αφορά τη βιωσιμότητα, την οικονομία και την υγεία. Δυστυχώ, αν κοιτάξουμε τις ε, παρούσε τάσεις, εάν ε, δεν πετύχουμε κάποιες αλλαγέ με τις πολιτικές μας και με καινοτομίε, η κατάσταση ε, δεν θα είναι καλή στο εγγύς μέλλον, ούτε όσον αφορά την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Χρειαζόμαστε, λοιπόν, πολιτική δράση και νέες τεχνολογίες για να αντιστρέψουμε τις τάσεις. στο Κοινό Κέντρο Ερευνών. Ε, διενεργούμε έρευνες και συνεργαζόμαστε με τα άλλα 30 τμήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, καλύπτουμε λοιπόν θέματα όπως είναι η μετανάστευση, οι μεταφορές, η ενέργεια, το περιβάλλον, ε, η γεωργία και η ασφάλεια. Όλοι αυτοί οι σε όλους αυτούς τους τομείς προσπαθήσαμε πέρσι ε, να εκπονήσουμε ε, εκθέσεις ε, εμβληματικές για να ενημερώνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις πιο σημαντικές τάσεις. Και εδώ στην αίθουσα θα βρείτε τις δημοσιεύσεις μας. Παρακαλώ λοιπόν να πάρτε ό,τι σας ενδιαφέρει. Είχαμε εκθέσεις ε, για κάποιες σημαντικές τεχνολογίες όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Ε, για το μέλλον των πόλεων είχαμε μια έκθεση για το μέλλον της εργασίας και τις δεξιότητες και υπάρχει και μια τέτοια έκθεση σχετικά με το μέλλον των οδικών μεταφορών. Θα σας περιγράψω τα σημαντικά σημεία της έκθεσης για το μέλλον των οδικών μεταφορών. Η έκθεση αυτή εξετάζει τις τεχνολογίες και τις κοινωνικές τάσεις ε, και εξετάζουν τι εξελίξεις θα έχουμε τα επόμενα 50 χρόνια. Τέσσερις ε, παράγοντες εξετάζουμε, αυτοματοποίηση, διασυνδεσμότητα, ε, τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξιδίων του άνθρακα και την οικονομία του διαμοιρασμού διότι θεωρούμε ότι αυτοί είναι οι τέσσερις σημαντικότεροι παράγοντες για τις οδικές μεταφορές στην Ευρώπη. Ε, προβλέπουμε λοιπόν τι εξελίξεις θα υπάρξουν ε, μέσα στην επόμενη δεκαετία. Στην επόμενη διαφάνεια θα σας δώσω κάποια παραδείγματα τέτοιων τάσεων. Γενικά, οι έρευνες δείχνουν ότι η διασυνδεσιμότητα και η αυτοματοποίηση μπορεί να αυξήσει ε, την ε, χωρητικότητα των ε, δρόμων κατά 80% και μπορεί να μειώσει κατά 90% τα ατυχήματα. Πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία αυτά λοιπόν. Ωστόσο, η αρνητική πλευρά είναι ότι μπορεί να αυξήσει την παρουσία αυτοκινήτων στους δρόμους μας. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, την, ε, ε, τις ε, μεταφορές του διαμοιρασμού. Έχουμε την Uber και την Lyft που είναι τα συστήματα που χρησιμοποιούνται περισσότερα. Βλέπουμε λοιπόν αύξηση της χρήσης των αυτοκινήτων διότι οι άνθρωποι δεν, παίρνουν τις, ε, δεν χρησιμοποιούν τις μαζικές μεταφορές, ε, προτιμούν ε, τα αυτοκίνητα. Υπάρχει λοιπόν ο κίνδυνος να αυξηθεί πάνω από 5% η ζήτηση για μεταφορές. Και μέχρι 30% μπορεί να είναι η απώλεια από τις μαζικές μεταφορές. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ένα μείγμα θετικών και αρνητικών παραγόντων που θα πρέπει να εξετάσουμε. Η διαμόρφωση της πολιτικής ε, θα πρέπει να ασχοληθεί με όλες αυτές ε, τις ε, προκλήσεις με ολιστικό τρόπο. Ενδιαφέρουσα οδός είναι τα λεγόμενα ζωντανά εργαστήρια, living labs. Μια από τις βασικές ετάσεις που διαπιστώσαμε είναι ότι πρέπει να γνωρίζουμε την συμπεριφορά των πολιτών και πρέπει να ε, δοκιμάσουμε σε πραγματικές συνθήκες ε, τις ε, τεχνολογίες μας. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιούμε πολύ περισσότερα τα λεγόμενα ζωντανά εργαστήρια, δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες δηλαδή, για να μπορούμε να παρέχουμε καλές λύσεις ε, σε όσους διαμορφώνουν την πολιτική. Ένα τέτοιο εργαστήριο ήταν στην Ίσπρα, σε μια από τις έδρες μας, όπου θελήσαμε ε, να ε, εξετάσουμε την, τις αυτοματοποιημένες μεταφορές, τις διαμερισμένες μεταφορές και θα δοκιμάσουμε τις διάφορες δυνατότητες και θα ήθελα να σας καλέσω να επισκεφτείτε την Ίσπρα και να δείτε τι κάνουμε εκεί και σε αυτό το ζωντανό μας εργαστήριο, αλλά να δείτε τι δοκιμές κάνουμε. Ε, και πώς συλλέγουμε στοιχεία σχετικά με αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μία από τις τάσεις που σας εξήγησα στην προηγούμενη διαφάνεια μας για τις εκθέσεις μας ε, ήταν οι έρευνες για την ε, διασυνδεσιμότητα και θα Ήθελα να σας δείξω στη διαφάνεια αυτή πώς οι τεχνολογίες έρευνας και καινοτομίας μπορούν να ε, παρακολουθούνται σε όλη την Ευρώπη σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά ε, θέλουμε να δούμε και ποιες είναι οι κορυφές τεχνολογίες μας ε, όσον αφορά τις επενδύσεις και τι θέση κατέχει η Ευρώπη σε αυτό το τοπίο. Με το σύστημα τρίμης λοιπόν που καταγράφει τις τάσεις ε, στις μεταφορές ε, και στις καινοτομίες, διαπιστώσαμε ότι βλέπουμε αύξηση στις τεχνολογίες ε, ηλεκτρισμού και υδρογόνου, αλλά ε, κυρίως έχουμε τις τεχνολογίες πιλωτηρίου, και στα ε, συστήματα διαμοιρασμού. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ποιο επενδύει πού για να δούμε τι θέση έχει η Ευρώπη στο παγκόσμιο τοπίο και να δούμε πού υπάρχουν μεγαλύτερε δυνατότητε καινοτομία. Επίσης ε, ενδιαφέρον ε, είναι ότι ε, η απορρόφηση των τεχνολογιών αυτών από την αγορά είναι ακόμα πολύ αργή. Παρότι λοιπόν έχουμε τις καινοτομίες, καθυστερεί ακόμη η υιοθέτηση των τεχνολογιών αυτών από τις αγορές στην ε, διαφάνεια αυτή. Θα ήθελα να σας δώσω ένα στιγμιότυπο του τι κάνουμε στο Κοινό Κέντρο Ερευνών ε, όσον αφορά την διαλειτουργικότητα ε, στην Ευρώπη. Είναι λοιπόν ένα κέντρο που εξετάζει τη διαλειτουργικότητα ηλεκτρονικών οχημάτων, των φορτιστών τους και την ενσωμάτωσή τους στο FES δίκτυο. Έχουμε λοιπόν ένα κέντρο δοκιμών στην Ίσπρα ε, και εξετάζουμε εδώ πώς ε, μπορεί να γίνει η μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Εάν επισκεφτείτε λοιπόν ε, την Ίσπρα θα μπορέσετε να δείτε από κοντά τις εργασίες μας. Άλλο παράδειγμα είναι κάτι που κάνουμε στην Φλωρεντία. Ε, χωρητική κατανομή της ε, ζήτησης ενέργειας ε, και τις ανάγκες υποδομών φόρτισης. Οι πληροφορίες αυτές θα βοηθήσουν τις αρχές της πόλης να καταγράψουν τις κινήσεις και τις ανάγκες φόρτισης και έτσι οι δημοτικές αρχές θα μπορέσουν να σχεδιάσουν τις υποδομές τους. Είναι λοιπόν πολύ σημαντική η χωροταξική ανάλυση και αποτελεί τμήμα των εργασιών μας. Αυτή η διαφάνεια δείχνει τι κάνουμε όσον αφορά τις μπαταρίες, τους συσσωρευτές. Συμμετέχουμε στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία Συσσωρευτών, ε, κάτι που ξεκίνησε η προηγούμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μελετάμε λοιπόν ε, την χρήση της τεχνολογίας και της τάσης για να στηρίξουμε τη διαμόρφωση πολιτικής στον τομέα αυτών. Οι αναλύσεις μας δείχνουν ε, ότι οι μπαταρίες λιθίου ιονίου θα γίνουν πιο οικονομικές λόγω της ανακύκλωσης των μπαταριών αυτών. Η ε, επανάχρηση και η ανακύκλωση μπορεί να γίνουν ε, για ε, χρήση στην ενέργεια και μετά, για παράδειγμα, το τέλος ζωής σε μια τέτοια μπαταρία αυτοκινήτου. Και βλέπετε εδώ στο δεύτερο στη δεύτερη ζώνη δεδομένων πόσο μπορεί να αυξηθεί αυτή όσον αφορά το μερίδιο της αγοράς. Και στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η Ευρώπη ε, κατέχει μόνο το 3% αυτού του τμήματος της αγοράς, ε, αλλά ε, πιστεύουμε ότι μέχρι 25% μπορεί να φτάσει το μερίδιο αυτό και να δημιουργήσουμε μια εσωτερική αλυσίδα αξία για τι μπαταρίε. Αυτό είναι κάτι που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Πιστεύουμε όμω ότι με τη συμμαχία θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε αυτή τη δυνατότητα. Η επόμενη διαφάνεια δείχνει τις ε, δραστηριότητες ε, δοκιμών σε συσσωρευτές ε, του Κοινού Κέντρου Ερευνών. Αφενός εξετάζουμε την αποδοτικότητα των μπαταριών που είναι σημαντικός παράγοντας για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Εξετάζουμε όμως και τα πρότυπα για την απόδοση των παταριών ε, για να μπορέσουμε να ε, στηρίξουμε τη βιωσιμότητα του τομέα. Διάφορες πτυχές λοιπόν όσον αφορά τις δοκιμές ε, μπαταριών, κάτι που μπορεί να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα ε, και την ε, εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Σας μίλησα για τα σημεία συμφόρησης στους δρόμους. Άλλη δουλειά που κάνουμε λοιπόν είναι οι δείκτες που χρησιμοποιούμε για να μπορέσουμε να μειώσουμε τη συμφόρηση. Βλέπετε εδώ ένα σχεδιάγραμμα που δείχνει τον μέσο χρόνο ανά έτος που περνούν οι οδηγοί μας ε, στην κίνηση. 40 ώρες το χρόνο για κάθε Ευρωπαίο ε, μία εβδομάδα, μία εργάσιμη εβδομάδα δηλαδή και μιλάμε μόνο για τη συμφόρηση. Όταν έχει σταματήσει, όταν έχει κολλήσει το αυτοκίνητο και παραμένει ακίνητο. 40 ε, ώρες το χρόνο είναι αυτό συνολικά. Και τελικές παρατηρήσεις όσον αφορά τις κοινωνικές συνέπειες ε, από την κινητικότητα. Είναι εργασίε που θα συνεχίσουμε και στο μέλλον. Εξετάζουμε λοιπόν πώ οι νέε τεχνολογίε και οι νέοι τρόποι μεταφορά επηρεάζουν ε, συνολικά την οικονομία και την απασχόληση. Ένα παράδειγμα, τα, ηλεκτρικά οχήματα περιέχουν μόνο 35 κινητά σημεία σε σχέση με τα 167 ε, στο ε, Volkswagen Golf, ε, στην μηχανή εσωτερικής καύσης του. Αυτό δείχνει ότι μάλλον ε, θα έχουμε πολύ λιγότερες θέσεις απασχόλησης ε, ως αποτέλεσμα ε, της κατασκευής των ηλεκτρικών οχημάτων. Ωστόσο, ο τομέας των συσσωρευτών από μόνο του και, και αν δημιουργήσουμε μια εσωτερική αλυσίδα αξίας για τις εταιρείες, για τις μπαταρίες, συγγνώμη, θα έχουμε δημιουργία περισσότερων θέσεων απασχόλησης. Αυτό λοιπόν είναι ένα παράδειγμα για το πόσο όλα αυτά θα επηρεάσουν την οικονομία. Κατόπιν, οι τελικέ μου παρατηρήσει, ε, τι μέλλον έχουν οι οδικέ μεταφορέ. Το δικό μα συμπέρασμα είναι ότι οι τεχνολογικέ αλλαγέ από μόνε του δεν θα μπορέσουν να μα δώσουν το μέλλον ε, στι μεταφορέ που θέλουμε. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε και δύο άλλε αλλαγέ. Το ένα είναι η διακυβέρνηση. Οι νέε τεχνολογίε θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ε, για να δημιουργηθούν, να αναπτυχθούν νέα πρότυπα διακυβέρνηση, ώστε να έχουμε καλύτερη κατανομή της κίνησης στους δρόμους ε, και να έχουμε ρυθμισμένη πρόσβαση στις οδικές υποδομές για να βελτιστοποιήσουμε τη χρήση τους ε, για όλα τα μέσα μεταφοράς. Και το δεύτερο σημείο που είναι ζωτικής σημασίας για μένα είναι ότι θα πρέπει να συνομιλούμε με τους πολίτες διότι αυτοί είναι οι βασικοί χρήστες των νέων τρόπων μεταφορών και εάν δεν συνεργαστούμε με τους πολίτες δεν θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε το μέλλον που θέλουμε η οικοδόμηση εμπιστοσύνη ε, περνάει μέσα από τη συνεργασία με τους πολίτες. Αυτά ήθελα να σας δώσω ω εισαγωγή. Εδώ βλέπετε τις, ε, τα στοιχεία της ε, ιστοσελίδα μας που μπορεί να σας ενδιαφέρει. Σας καλώ όμω να έρθετε στην Ίσπρα και να δείτε από κοντά τις αναλυτικές και εργασιακέ μας εργασίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Äh, Κυρία Βιτσέβα, σας ευχαριστώ πολύ για την ε, εισήγησή σας. Ε, πολύ ευχαρίστω θα ανταποκριθούμε στην πρόσκλησή σας ε, να πάμε στην Ίσπρα. Ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Έπασε τόση πλάκα κάνω. δύο πολύ ενδιαφέροντα θέματα έχουμε σήμερα λοιπόν στην ημερήσια διάταξη. και θα ε, λάβετε σύντομα και τις ερωτήσεις μας. Ε, πάλι λοιπόν θα ακούσουμε πρώτα τους ε, εισηγητές των πολιτικών ομάδων. Από το ΕΛΚ ο συνάδελφος Σαλίνη θα θέσει ερώτηση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Μου άρεσε πάρα πολύ η παρουσίαση για διάφορους λόγους. Είναι σαφές ότι όταν μιλάμε για έρευνα και καινοτομία, εμείς έχουμε μια ανησυχία. Και αυτό οφείλεται στη συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή για τον προπολογισμό. Ξέρετε πολύ καλά, όλο το κομμάτι που συνδέεται με την έρευνα και καινοτομία μας δημιουργεί πάρα πολύ πρόβλημα λόγω των προτάσεων που έχουν κατατεθεί. Έχουμε μπλέξει αυτή τη συζήτηση, έχει γίνει λαφυρινθόδηση συζήτηση και νομίζω ότι με βάση προτάσεις προβλέπεται περαιτέρω μείωση 30% για την έρευνα ε, και 3% ε, σε σχέση με την αρχική πρόταση της Κομισιόν για τον ορίζοντα. Είναι ένα στοιχείο που πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Έχω και ένα συγκεκριμένο όμως θέμα που θέλω να θίξω, που πάντα με ενδιαφέρει όταν μιλάμε για τον ορίζοντα. Εγώ είχα κάποια προβλήματα για αυτή την ε, κατανομία ανακλάστερ σε σχέση με το παρελθόν στο παρελθόν δεν υπήρχε. Κάποια προβλήματα τα έχω ε, γιατί διαρωτώ με πώς δημιουργήθηκαν καταρχάς αυτά τα κλάστερ. Ε, οι μεταφορές και η κινητικότητα δεν μπαίνουν μαζί με την βιομηχανία, μπαίνουν μαζί με το κλίμα. Η απάντηση είναι προφανής. Οι μεταφορές είναι στο κέντρο της προσοχής όλων και είναι ο βασικός κατηγορούμενος για τη μόλυνση. Εντάξει, αλήθεια είναι, αλλά από την άλλη είναι αλήθεια ότι έχουν και άλλη χρησιμότητα οι μεταφορέ. Πέρα από του κινδύνου δηλαδή που προκαλούν, έχουν και άλλη χρησιμότητα. Και έχω πρόβλημα που του κολλήσαμε, που του χώσαμε και που του χώσαμε τι τις μεταφορές. Ε, επίσης, μιλάμε για αυτοματοποίηση, ε, συνδεσιμότητα και αυτό ε, συνδέεται φυσικά με την πραγματική χρήση και ωφέλεια των μεταφορών. Εμείς εδώ, στο εσωτερικό του Κοινοβουλίου, όταν μιλάμε για τις μεταφορές, 9 στις 10 φορές μιλάμε για την μείωση των εκπομπών διοξείδου του άνθρακα. Ποτέ δεν μιλάμε ή πολύ λίγο μιλάμε, εν για την αυτοματοποίηση και τα λοιπά, την συνδεσιμότητα και τα λοιπά. Επομένως, είναι ευθέο να γίνει μια εντατικοποίηση της ε, ερευνητική προσπάθειας που συνδέεται με την προστιθέμενη αξία των μοντέρνων μεταφορών ε, μέσα σε ένα νέο πλαίσιο και μοντέλο ανάπτυξης που θέλουμε να προτείνουμε. Πολύ ωραία. Με βάση όλα αυτά που σας είπα, σας ρωτάω, κατά την άποψή σας, εσείς που κάνατε την πολιτική συζήτηση που κάναμε τώρα την, ε, σε αυτό το χώρο, τι κίνδυνο πιστεύετε ότι ε, μπορεί να μας δημιουργήσει αυτή η εμπάθεια που έχουμε στη συζήτηση ε, και η μονομανία που έχουμε αναπτύξει συζητώντας την ε, μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ντάνιελσον από το S&D. Ε... Ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ για την παρουσίαση. Άκουσα περισσότερα και έμαθα περισσότερα για τη δουλειά σα. ενδιαφέρονταν αυτό. Είδα τι δυσκολίε, αλλά και τις, τη σημασία του τομέα των μεταφορών για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω λίγε ερωτήσει. Εγώ όμω θα εστιάσω βεβαίω στο θέμα τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Η έρευνά σας εστίασε στην, στα ηλεκτρικά οχήματα, αλλά θα μπορούσατε να πείτε και δύο λόγια για τα εναλλακτικά καύσιμα και την άποψή σας για την πιθανή παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων και το πόσο μπορούν να αναπτυχθούν και να χρησιμοποιηθούν από διάφορους τρόπους μεταφορών. Υπάρχουν δυνατότητες, ας πούμε, για εναλλακτικά καύσιμα στις χερσαίες μεταφορές ή θα πάνε σε άλλους τομείς, ας πούμε, κατά προτεραιότητα τα εναλλακτικά, τα καύσιμα. Και για την ηλεκτροδότηση, τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας. Ε, για τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε ε, ηλεκτρική ενέργεια για μεγάλες μεταφορές. Γιατί υπάρχουν μεικτά μηνύματα. Δεν ξέρω αν μπορούμε, ας πούμε, να κινήσουμε ηλεκτρικά αυτά τα οχήματα που έχουμε σήμερα. Και αν όχι, θα μπορούσαμε ε, τουλάχιστον να χρησιμοποιήσουμε την ηλεκτρική ενέργεια, ας πούμε, σε ένα μεγάλο κομμάτι των χερσαίων μεταφορών, ας πούμε, και όταν βγαίνουν να, να μπορούν ας πούμε, να εφοδιάζονται σε, σε ηλεκτρική ενέργεια, να υπάρχει δυνατότητα ηλεκτροδότηση σε κεντρικού άξονε και όταν βγαίνουν εκτό να χρησιμοποιούν την μπαταρία. ευχαριστώ από το Ρηνιού, κύριο Φλέγκο. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την ομιλήτρια που μας παρουσίασε αυτό τα, αυτά τα πολύ σημαντικά στοιχεία. Εκ μέρους ε, των συντονιστών του Renew, έχω την τιμή να σας κάνω εγώ κάποιες ερωτήσεις. Χαίρομαι που μπορώ να σας θέσω αυτές τις ερωτήσεις, γιατί εγώ έχω πτυχίο ακριβώς για αυτά τα θέματα. Έχω σπουδάσει αυτά τα θέματα. Οι παρουσιάσεις σας, οι εκθέσεις σας είναι πολύ ψηλής ποιότητας και πολύ ενδιαφέρουσες και οι δημοσίευσεις σας. Τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει όλο και περισσότερη τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την αυτοματοποιημένη κίνηση. Έχουμε φτάσει σε τεχνολογία τρίτης γενιάς. Μιλάω για την αυτοματοποίηση. Για την τέταρτη γενιά τέτοιας τεχνολογίας αρχίζουμε να μιλάμε σιγά σιγά. Αλλά πότε νομίζετε ότι μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τους δρόμους για αυτά τα αυτόματα οχήματα. Τώρα θέλω να ρωτήσω κάτι για την ιεραρχία σας, για τους ανώτερούς σας. Οι ανώτεροί σας, επίτροποι, ακόμα και πρόεδρος επιτροπής, ενώ τι είδου ε, νομοθετήματα περιμένετε να υποβληθούν. Ξέρω ότι υπάρχουν θέματα προπολογισμού, αλλά εμένα με ενδιαφέρει τι κανονισμός, την νομοθεσία χρειάζεται, ούτως ώστε οι μεταφορές να γίνουν πιο πράσινες, να έχουμε αυτόματα οχήματα και να έχουμε την τέταρτη γενιά τεχνολογίας αυτοματοποίησης. Πότε θα είναι λειτουργική αυτή η τεχνολογία. Πότε θα την έχουμε στα χέρια μας. Επίσης θα ήθελα να κάνω και μια άλλη παρατήρηση. Να σας την πω και αν κάνω κάπου λάθος, διορθώστε με. Αν, Φερρυπίν, μπορούσαμε οι μισές μας πόλεις να χρησιμοποιούν μόνο ηλεκτρικά οχήματα, αυτό θα δημιουργούσε προβλήματα με, την, με τον ανεφοδιασμό σε ηλεκτρική ενέργεια αυτών των πόλεων. Υπήρχε περίπτωση να έχουμε ε, διακοπή ηλεκτρικού, ας πούμε, σε αυτές τις πόλεις. Ευχαριστούμε τον κύριο Φλέγκο. Από το ID. Συγγνώμη, από τους πράσινους η κυρία Πάουλους. Ευχαριστώ που ήρθατε και μας παρουσιάσατε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα, θα την κοιτάξω πιο λεπτομερό στο ίντερνετ, γιατί είναι πολύ καλή ποιότητα και μου άρεσε το γεγονό ότι έχετε διαφορετική προσέγγιση. Λέτε ότι θέλουμε κινητικότητα για, το... για του πολίτε, όχι για τα αυτοκίνητα. Γιατί στη Γερμανία και σε άλλε χώρε βλέπουμε ότι οι πόλει λένε. Θέλουμε να μας δοθεί πίσω ο δημόσιος χώρος, να δοθεί δηλαδή στους πολίτες. Ακόμα και οι άνθρωποι που, παρουσ... παραπονιούνται για την ε, κυκλοφοριακή του συμφόρηση ε, και που κολλάνε κάθε πρωί στα αυτοκίνητά τους λένε ε, ότι θέλουν περισσότερους δρόμους. Ε, αυτοί οι ίδιοι όταν πάνε ας πούμε σε άλλες πόλεις, στην Κοπενχάγη, λένε «Α, τι ωραία που είναι εκεί, ας πούμε, έχουν περισσότερα ποδήλατα και περισσότερο χώρο έχουν οι πεζοί, πούμε, και δεν συνειδητοποιούν ότι αυτά τα πράγματα είναι αλληλένδετα. Επίσης, θα μπορούσε να κάνει συγκεκριμένε προτάσει πολιτική, ούτω ώστε η Κομισιόν να έχει στα χέρια της καλή βάση έρευνα, δηλαδή, για να παρουσιάσει νομοθεσία για τους πολίτες. Επίσης, τι γίνεται ε, με τις περιοχές της Υπέθρου που δεν έχουμε τις ίδιες δυνατότητε για δημόσιες μεταφορές, γίνεται έρευνα για την κινητικότητα σε αυτές τις περιοχές ή κινητικότητα, ας πούμε, ανάλογα με τη ζήτηση. Εκεί όπου οι δημόσιες μεταφορές ε, δεν είναι τόσο τακτικές, γιατί είναι πολύ ακριβές, ας πούμε, για μικρούς δήμους και κοινότητες ή για χωριά, Φερρυπίν. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταίος συντονιστής από την ΚΟΕ, κυρία Κουντουρά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου για την ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας και θα ήθελα να ρωτήσω αν το Κοινό Κέντρο Ερευνών σκοπεύει να ασχοληθεί με το ζήτημα της κοινωνικά δίκαιης μετάβασης στον τομέα των μεταφορών. Είναι πολύ σημαντικό να εξετάσουμε σε ποιο βαθμό η μετάβαση θα επηρεάσει τους κοινωνικά πιο ευάλωτους αλλά και τους γεωγραφικά πιο ευάλωτους όπως είναι τα νησιά και οι απομονωμένες περιοχές της Ευρώπης για να προτείνουμε βέβαια τα απαραίτητα αντίμετρα. Επίσης, έχετε μελετήσει αρκετά το ζήτημα των εναλλακτικών καυσίμων που μας απασχολεί και μας ιδιαίτερα στην Επιτροπή μας, την Επιτροπή Τραν. Θα σταθώ στο υδρογόνο, το οποίο όπως μας είπατε απορροφά μεγάλο ποσοστό των επενδύσεων στις μεταφορές και το οποίο φαίνεται να υπόσχεται πολλά για τη βιωσιμότητα των μεταφορών. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε τη γνώμη σας για το πότε μπορεί αυτή η τεχνολογία να γίνει ανταγωνιστική, υπό ποιε προϋποθέσεις, τόσο για τις οδικές μεταφορές, τις θαλάσσιες μεταφορές, αλλά ακόμα και για τις αεροπορικές μεταφορές και σε ποιο ποσοστό πιστεύετε ότι μπορεί το υδρογόνο να αντικαταστήσει τα συμβατικά καύσιμα. Ευχαριστώ πολύ. Vielen Dank. Jetzt haben wir noch aus den Reihen der Abgeordneten zwei weitere Fragen. Άλλες δύο ερωτήσει έχουμε από ευρωβουλευτές. Ε, την κυρία Τάλερ καταρχάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Βιτσέβα για την παρουσίασή σας. Πράγματι, πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία που ακούσαμε και σας συγχαίρω και για τις εμβληματικέ εκθέσεις ε, που αναφέρατε. Δύο σύντομες ερωτήσεις έχω. Η πρώτη έχει να κάνει με ε, την διαφορά στην κινητικότητα στις ε, πόλεις και στην Ήπεθρο, στις αγροτικές περιοχές. Ε, μας είπατε ότι 40 ώρες το χρόνο ε, κολλάμε στην κίνηση και ότι αυτό έχει και αρνητικές οικονομικές συνέπειες και 1 έως 2% πόλεις. Αυτό είναι ο μέσο όρο στο σύνολο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, εξετάσατε αν υπάρχουν διαφορέ ανάμεσα στι ε, αστικέ ε, και αγροτικέ περιοχέ, η πρώτη μου ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση για τι μπαταρίε. Συχνά όταν μιλάμε για ηλεκτρικά οχήματα, ακούγεται, ακούγονται αμέσως αρνητικά ε, λόγια για τις μπαταρίες, ε, τι κάνουμε για παράδειγμα ε, σε περίπτωση ατυχήματος. Έχετε πρωτοβουλίες δεύτερης ζωής, έχετε εξετάσει τα ενδεχόμενα δεύτερης ζωής για τις μπαταρίες αυτές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχω και εγώ μια ερώτηση την οποία θα ήθελα να σας θέσω. λίγο προς την κατεύθυνση της ερώτησης της κυρίας Τάλερ για τις ε, μπαταρίες στα ηλεκτρικά οχήματα. Μια από τις ε, μεγαλύτερες ε, προκλήσεις θα είναι όταν δεν είναι πια χρήσιμη για το όχημα η μπαταρία αυτή. Όταν έχει πέσει η απόδοση στο 80% θα πρέπει να αλλάχτεί η μπαταρία. Θα πρέπει να ανακυκλωθεί λοιπόν αλλά από ό,τι μου λένε οι εμπειρογνώμονες ε, υπάρχει ένα βήμα πριν που πρέπει ε, να εξετάσουμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την μπαταρία αυτή ως ε, αποθήκη ενέργειας. Εάν θέλουμε να αναπτύξουμε περαιτέρω τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ηλιακή ή την αιωλική, θα πρέπει να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τις ε, δυνατότητες αποθήκευσης ε, κατά τις ώρες εχμής, ε, το μεσημέρι για την ηλιακή ενέργεια για παράδειγμα. και ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν οι μπαταρίες αυτές έχει υποθεί. Έχετε σκεφτεί πώς μπορεί να γίνει αυτή η δεύτερη χρήση των μπαταριών διότι περιέχουν ε, πολύ σημαντικά και σπάνια υλικά και επίσης ε, πώς μπορούν να ανακυκλωθούν. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω όλους για την θετική ανταπόκριση στις εργασίες του Κοινού Κέντρου Ερευνών. Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι πρέπει να πω ότι το κέντρο μας κάνει έρευνα μόνο. Δεν είμαστε εμείς εκείνοι που προτείνουμε πολιτικές. Εμείς υποστηρίζουμε την υιοθέτηση πολιτικών τις οποίες αναπτύσσουν οι συνάδελφοι από τις αντίστοιχες μονάδες πολιτικής στα διάφορα τμήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επομένως, εγώ θα είμαι πάρα πολύ προσεκτική να μην βγω έξω από τα χωράφια μου και είναι πάρα πολύ ευαίσθητο αυτό. Ε, είναι πολύ σημαντικό το Κοινό Κέντρο Ερευνών να παραμένει ουδέτερο σε σχέση με τις πολιτικές επιλογές ε, αυτό είναι απαραίτητο για να ε, παραμένει η εμπιστοσύνη σε εμά. Επομένω, οποτεδήποτε με ρωτάτε τη μία ή την άλλη επιλογή πολιτική προτιμάτε, ή αν πιστεύετε ότι χρειάζεται ρύθμιση στον τάδε τομέα, θα είμαι πολύ προσεκτική στο τι θα απαντήσω για να μην εκφράσω προσωπικέ απόψει σαν να ήταν του κέντρου. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το ζήτημα του προπολογισμού. Σήμερα είναι η πιο σημαντική ημέρα. Ελπίζω ε, πραγματικά να υπάρξει συμφωνία πρώτα απ' όλα, γιατί κάτι τέτοιο θα καταδείξει ότι η Ευρώπη είναι σε θέση να λαμβάνει αποθέσει. και πραγματικά πιστεύω να συμφωνήσουν οι ηγέτε των κρατών σε έναν σωστό αξιοπρεπή προπολογισμό. Φυσικά δεν μπορώ να κάνω κάποιο σχόλιο αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή η απόφαση είναι στα χέρια των αρχηγών των κρατών μελών να λάβουν μια ουσιαστικά υπεύθυνη απόφαση. Μιλήσατε για το νέο πρόγραμμα Horizon Europe. Ε, και πάλι αυτό δεν είναι αρμόδιότητα του κέντρου, είναι της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας. Οποτεδήποτε υπάρχει σύνδεση των μεταφορών με τη, των, τις προσπάθειες για το κλίμα, έχουμε μια συγκεκριμένη ομάδα για διεύθυνση για την ε, σχέση των μεταφορών και της ενέργειας με το κλίμα, βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν σχετίζεται και η συμμετοχή της βιομηχανίας. Επομένως θα πρέπει να αναμείνουμε, να δούμε την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βιομηχανική στρατηγική που θα γίνει στις 10 Μαρτίου. Επομένως οτιδήποτε αναφέρεται στον παραγωγικό τομέα θα το βρούμε σε αυτή την πρόταση. Εάν βεβαίως συνδέεται με το κλίμα και με την απεξάρτηση από τον άνθρακα δεν σημαίνει ότι δεν θα συμπεριλάβουμε ή δεν θα θεωρήσουμε και τον τομέα των μεταφορών ως έναν τομέα στον οποίο να μπορούν να αναλυφθούν παραγωγικές πρωτοβουλίες. Ο στόχος είναι μέχρι το 2050 να είμαστε ουδέτεροι από πλευράς α, χρήσεως άνθρακα. Αυτό στην Ευρώπη είναι κάτι που δημιουργεί ψηλού επίπεδου ε, απαιτήσει ε, και σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα θα χρειαστεί να έχουμε και μια ομάδα πρωτοβουλειών, ένα κλάστερ πρωτοβουλίων για την εξάρτηση από τον άνθρακα. Αναφέρομαι προφανώ στην κινητικότητα. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι έχει ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία ο τομέα των μεταφορών γιατί είναι ο τομέας ο οποίος συνδέει τους υπόλοιπου τομεί της οικονομίας μεταξύ τους. Επομένω, ο τομέας των μεταφορών είναι πολύ σημαντικός. Για τα εναλλακτικά καύσιμα θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο που είναι ειδικό για να σας δώσει πολύ πιο συγκεκριμένες και εξειδικευμένες απαντήσεις. Ε, Πράγματι, ε, εργαζόμαστε πολύ στο θέμα του υδρογόνου και για να απαντήσω στις ερωτήσεις σας τις σχετικές. Ξέρετε ότι στο πλαίσιο του ορίζοντα 2020 υπήρχε μια κοινή πρωτοβουλία για την χρήση του υδρογόνου. Και κατά τη διάρκεια αυτών των πέντε ετών, κάτι λιγότερο από πέντε χρόνια, σχεδόν πέντε χρόνια λοιπόν που είχαμε αυτή την κοινή πρωτοβουλία, κοινό εγχείρημα, υπήρξε συνεργασία μεταξύ ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων για να αναπτυχθούν τέτοιες τεχνολογίες. Το κόστος της χρήσης του υδρογόνου μειώθηκε κατά πολύ. Και θα έλεγα ότι έχουμε ήδη φτάσει πολύ κοντά στο να είναι το κόστος του πραγματικά ανταγωνιστικό με άλλα ε, άλλους, άλλες πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται στον τομέα των μεταφορών. Επομένως, ε, έχουμε ήδη λεωφορεία στόλους λεωφορείων που κινούνται με υδρογόνο. Έχουν γίνει πολλές σημαντικές πρόοδοι τα τελευταία πέντε χρόνια ε, και στη μείωση του κόστους αλλά επίσης και στη βελτίωση της ασφάλειας. Θα συνεχιστεί αυτή, αυτό το κοινό εγχείρημα. Πιστεύω πως ναι. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών συμμετέχει σε αυτό το κοινό εγχείρημα και συμβάλλει με τις ερευνητικές του εργασίες. Για το ζήτημα τώρα του εξηλεκτρισμού και πιο συγκεκριμένα αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ηλεκτρική ενέργεια για τις μεταφορές μεγάλων αποστάσεων, εάν υπάρχουν κάποιες εναλλακτικέ για να χρησιμοποιηθούν οι υποδομές του δικτύου και πάλι θα τα αναθέσω αυτά να τα απαντήσει καλύτερα ο ειδικό συνάδελφος. Τώρα, για το ζήτημα του αυτοματοποίησης και της λεγόμενης τέταρτης γενιάς, όσον αφορά τις πόλεις. Εγώ θα ήθελα να σας ζητήσω να, διαβάσετε την έκθεση που εκδώσαμε για τις, το μέλλον των πόλεων, γιατί αναφερόμαστε και στον τομέα των μεταφορών στο εσωτερικό της πόλης. Επίσης, αναφερόμαστε στο πώς, στη χωροταξία ε, σε μια πόλη, κατά πόσον είναι επισκόπημο ένας χώρος να χρησιμοποιηθεί για οδούς ή για κάτι άλλο. Και αυτή τη στιγμή εμείς ε, αντιμετωπίζουμε την κινητικότητα ως μια υπηρεσία δεν το κοιτούμε υπό το πρίσμα των αυτοκινήτων ή από το πρίσμα μιας συγκεκριμένης μεθόδου, αλλά το βλέπουμε σαν μια υπηρεσία και κοιτούμε πώς μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματική ως υπηρεσία. Αυτό θεωρούμε ότι είναι η σωστή προσέγγιση. Δεν είναι ε, κάτι που σχετίζεται μόνο ή αποκλειστικά με τα αυτοκίνητα, το στόλους ή τις υποδομές. Ο στόχος θα πρέπει να είναι πώς μπορούμε να παράσχουμε αυτή την υπηρεσία όσο πιο καλά μπορούμε. Έτσι, σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να βλέπουμε την κινητικότητα. Τώρα για τις αγροτικές περιοχές, σε μία από τις διαφάνειες που σας έδειξα, ε, είδατε ότι έχουμε περίπου 40 ώρες το χρόνο ε, να σπαταλώνται από τους πολίτες της Ένωσης σε μποτιλιαρίσματα. Θα δείτε ότι υπάρχει μία μείωση από χώρα σε χώρα και ότι οι χαμηλότερες αυτές τιμές ε, τις ε, παρατηρούνται ε, στις μη περιοχές. Την έχουμε ήδη κάνει λοιπόν αυτή την ανάλυση για τη συμφόρηση και έχουμε επίσης και κάποιες συγκεκριμένες μελέτες που δεν αναφέρονται στη συμφόρηση μόνο στο, στις πόλεις αλλά και σε μη αστικές ή περιαστικές περιοχές. Τώρα, αυτό που θα ήταν πολύ χρήσιμο να γνωρίσω από τη δική σα την πλευρά είναι, ποια είναι το, ποια είναι, σε, σε ποιους τομείς λείπει η πληροφόρηση, λείπει η γνώση και πώς θα μπορούσαμε εμείς ω κοινό, κοινό κέντρο ερευνών ή και σε συνεργασία με άλλα ερευνητικά κέντρα να καλύψουμε αυτό το χάσμα, αυτό το κενό. Να ξέρουμε δηλαδή ποιε πληροφορίε και γνώσει σα λείπουν για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τι πολιτικέ συζητήσει που θα κάνετε από εκεί και πέρα. Ε, αν μπορείτε να εντοπίσετε οποιοδήποτε τέτοιο κενό, σα προσκαλώ να μα ενημερώσετε. Τώρα, μια μελέτη για την δίκαιη μετάβαση, με ρωτήσατε. Πράγματι, είναι ένα τομέα στον οποίο ε, έχουμε εργαστεί. Ε, κάναμε μια πιλωτική έναρξη ε, μια πρωτοβουλία ειδικά για τις περιοχές οι οποίες, ε, στις οποίες γίνεται εξόριξη άνθρακα και θα πρέπει να μεταβούν για να δούμε ειδικά σε αυτές τις περιοχές τι κοινωνικές επιπτώσεις θα έχει αυτή η μετάβαση. Έχουμε ήδη λοιπόν μια σχετική έκθεση ως παράδειγμα, μπορείτε να τη δείτε, ε, για να δείτε τι κάναμε στον τομέα αυτό θα συνεργαστούμε επίση με τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακή Ανάπτυξη, τη Regio, η οποία θα έχει στη διάθεσή τη τα 5,2 δισεκατομμύρια του Ταμείου Δίκαιη Μετάβαση και θα παράσουμε πληροφορίε και γνώση προ αυτήν. Προς αυτήν. Έχουμε λοιπόν ήδη δραστηριοποιηθεί στον τομέα αυτό και θα κάνουμε και πολλά παραπάνω. Τώρα για την δεύτερη ζωή που μπορεί να έχει μια μπαταρία σας το παρουσίασε ήδη, είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς μπορεί να επαναχρησιμοποιηθούν οι μπαταρίες, ιδίω εάν μιλούμε για τις πρώτες ύλε που έχουν χρησιμοποιηθεί και είναι στο εσωτερικό αυτών των συσσωρευτών. Πώς μπορούμε δηλαδή σε δεύτερη φάση να ξαναχρησιμοποιήσουμε αυτά τα υλικά. Πράγματι, μία εφαρμογή είναι να χρησιμοποιείται για αποθήκευση ενέργειας. Ε, μια ιδέα, μια, ένα ενδεχόμενο είναι να χρησιμοποιείτε μια μπαταρία αυτοκινήτου, ηλεκτρικού αυτοκινήτου, αφού εκπνεύσει η ζωή του στο αυτοκίνητο, να χρησιμοποιείτε οικιακά, να την φορτίζει κανείς το βράδυ και να τον χρησιμοποιεί ε, το πρωί ή να τη χρησιμοποιεί αν δεν χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο. Για εμάς το σημαντικό είναι να έχουμε μια ευφυή χρήση όλων των δυνατοτήτων αποθήκευσης ενέργειας που έχουμε διαθέσιμες. Και αν τελικά αυτά τα αυτοκίνητα, τα ηλεκτρικά, ε, αντικαταστήσουν σε μεγάλη κλίμακα τα παραδοσιακά, τα συμβατικά, σημαίνει ότι θα έχουμε στη διάθεσή μας μια μεγάλη δεξαμενή και δυνατότητα μάλλον αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτά από την πλευρά μου, τώρα μου θα δώσω το λόγο στον εξειδικευμένο τώρα συνάδελφο για να απαντήσει πιο συγκεκριμένα σε κάποιες από τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να, δώσω, να δώσω απάντηση σε τα θέματα ηλεκτροδότησης, εναλλακτικά καύσιμα. Τι γίνεται όταν έχουμε πιο περίπλοκους τομείς μεταφορών, όπως παραδείγματο χάρη ε, τις θαλάσσιες μεταφορές, τις μεταφορέ μεταφορές ε, αγαθών. Υπάρχουν απόψεις για αυτά τα θέματα. Αλλά εμείς είμαστε επιστήμονες πάνω απ' όλα. Δεν εκφράζουμε απλώς απόψεις και δεν προτάσουμε απόψεις. Θα το ξέρετε ίσως ότι δεν υπάρχει μία λύση για όλα. Υπάρχουν διαφορετικές λύσεις που εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες και θα πρέπει να βρούμε ποιε είναι αυτές οι κατάλληλες λύσεις. Ε, στον τομέα των μεταφορών έχουμε διάφορες δυνατότητε για μεταφορά ή αποθήκευση ενέργεια. Δεδομένων των στόχων για μια που έχουμε για το 2050 για μια κοινωνία α, ουδετέρων μεταφορών, πρέπει να ξεκινήσουμε τις συζητήσεις με τη Γενική Διεύθυνση Κλίματος για την αναθεώρηση των στόχων εκπομπών διοξείου του άνθρακα στις χερσαίες μεταφορές και θα πρέπει να κοιτάξουμε όλες τις λεπτομέρειες για το τι υπάρχει στην αγορά, τι υπάρχουν, τι τεχνολογίες υπάρχουν, τι καύσιμα έχουμε και πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε καλύτερα στις μεταφορές. Για την εκδοδότηση των φορτηγών Υπάρχει δυνατότητα να το κάνουμε, αλλά πέρα από κάποιες δοκιμές που έχουμε κάνει με φορτηγά σε κάποια κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν βλέπουμε μία ανάπτυξη σε μεγάλη κλίμακα τέτοιων φορτηγών. Όταν δείτε το κόστος των υποδομών, καταλαβαίνετε ότι η ηλεκτροδότηση όλων, ας πούμε, των αυτοκινητοδρόμων επισύρει ένα τεράστιο κόστος πέρα από τις ε, δυσκολίες που έχει η ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας. Θα θέλουμε γραμμές, ας πούμε, ε, ηλεκτρικής ενέργειας ε, στα τούνελ, στις γέφυρες, παντού. Για τα βαρέα οχήματα έχουμε διάφορες εναλλακτικές. Έχουμε τα βιοκάψιμα ή εναλλακτικά καύσιμα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Καθώς και για τις εσωτερικές, την εσωτερική ναυσιπλοεία, υγροποιημένο φυσικό αέριο. Για τομέα της αεροπορίας τώρα. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Έχουμε ε, κυψέλες υδρογόνου, αλλά δεν μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε στην αεροπλο... Ε, αεροπλοεία. Γιατί για να κουβαλάει το αεροσκάφος ε, τέτοιες ε, κυψέλες υδρογόνου έχουν τέτοιο βάρος που δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να πάμε προς αυτή τη λύση. Θέλουμε μεγαλύτερη καινοτομία. Γιατί όταν υπάρχει ανάγκη και υπάρχει και αγορά, κάποιο τελικά θα βρει τη λύση και θα την αναπτύξει. Για το υδρογόνο, για τις κυψέλες υδρογόνου, έχουμε κατασκευαστές που αναπτύσσουν τέτοια τεχνολογία και για τα και για τις μεταφορές μέσω βαρέων οχημάτων και για τα γεωταχή. Έχουμε δύο κυψέλες ε, στα βαρέα οχήματα, δηλαδή αντί για μία κυψέλη που έχουμε στα ελαφρά οχήματα. Αλλά δεν αποφασίζει η έρευνα για αυτά, είναι η αγορά που αποφασίζει και αυτή που θα βρει την καλύτερη και την πιο αποτελεσματική σε σχέση με το κόστος λύση. Νομίζω ότι τα κάλυψα όλα τα στοιχεία όλες τις ερωτήσεις που ακούστηκαν και αν όχι, βεβαίως, εδώ είμαι. Ξαναρωτήστε. Vielen Dank für die Stellungnahme. Wir werden mit Sicherheit σας ευχαριστώ πολύ. Σίγουρα θα έχουμε πρόσθετες ερωτήσεις, όχι σήμερα όμως, διότι ολοκληρώσαμε τη σημερινή συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Ευχαριστώ τους Ευρωβουλευτές, τη Γραμματεία, τους Διερμηνείς, λέει ο Πρόεδρος και εμείς ευχαριστούμε. Ε, στις 16 και 17 Μαρτίου πάντως θα ξαναβρεθούμε, όποιος έχει όρεξη, ε, να έρθει εδώ στην Επιτροπή Μεταφορών. Λήξη λοιπόν της συνεδρίασης. Καλή επιστροφή εύχομαι σε όλους ε, και καλό Σαββατοκύριακο.